Alors, euh, chers collègues, avant de... Πρωτού δώσω το λόγο στην κυρία Τσόρτσεβα, αγαπητοί συνάδελφοι, Σα υπενθυμίζω ότι το σημείο 18, σημείο 18, προθεσμία τροπολογιών είναι 26 Μαΐου το μεσημέρι ή τι αύριο το μεσημέρι. Και πάμε σε ένα πολύ σημαντικό σημείο στην μέση διαταξή μα την παρουσίαση των προτεραιοτήτων για την ανθρωπιστική βοήθεια του 2012 και χαίρομαι που μπορώ και πάλι να υποδεχτώ στην Επιτροπή μας την κυρία Κρυσταλίνα Τζόρτζεβα που είναι η Αρμόδια και το αντικείμενο της συζήτησής μας είναι ο διαρθρωμένος διάλογος για το έργο της Κομισιόν το 2012 δημόσια στο Συμφωνία Πλαίσιο που υπεγράφει μεταξύ Κομισιόν και Κοινοβουλίου τον Οκτώβριο του 2010 επιτρέπει στις κοινοβουλευτικές επιτροπές να συνεισφέρουν ιδέες για τις πρωτοβουλίε που θα θέλαν να δουν να ευδοκιμούν, μάλλον να αναλυθούν από την Κομισιόν το επόμενο έτος. Η Κομισιόν δεν έχει θεσπίσει ακόμα πρόγραμμα εργασία για το 2012, οπότε είναι η πρόσφορη και κατάλληλη στιγμή να συζητήσουμε με την Επίτροπο κυρία Τζόρτζεβα τους τομείς στους οποίους θα πρέπει να δώσει έμφαση η Κομισιόν του χρόνου. Μετά από το τέλος της συνεδρίασής μας σήμερα το απόγευμα, οι συντονιστέ θα αντλήσουν συμπεράσματα από τη συζήτηση με την κυρία Τσόρτζεβα και θα αποφασίσουν για τις, προτάσει προτάσεις που θα αποστείλουν στη συνέλευση των Προέδρων των Επιτροπών του Κοινοβουλίου για το πρόγραμμα της Κομισιόν του 2012 άνευ χρονοτριβής και κολυσιεργίας δυνατού λόγου στην κυρία Τζότζεβα. Έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε έντιμα μέλη του Κοινοβουλίου, κυρίες και κύριοι, χαίρομαι που μπορώ να επιστρέψω στην Επιτροπή Ανάπτυξη σήμερα. Οι ανταλλαγές απόψεων μέχρι τώρα με έχουν πείσει ότι μπορώ πάντα να βασίζομαι στα θετικά και επικοδομητικά σας σχόλια. Από τον Οκτώβριο που ήρθα για τελευταία φορά ενώπιον της Επιτροπής σας έχουμε δει να υπάρχουν μεγάλες αναστατώσεις στον αραβικό κόσμο, αλλά αντιμετωπίσαμε και μεγάλες καταστροφές, η κρίση στη Λιβύη, η κρίση στην ακτή του Αλεφαντοστού, η πολλαπλή κρίση της Ιαπωνίας και εξακολουθούν να υπάρχουν ακόμα συγκρούσεις και κρίσεις που συνεχίζονται στο Σουδάν, στη Μέση Ανατολή, στην δημοκρατική, δημοκρατία του Κονγκό και όλες αυτές οι καταστροφές και οι έκτακτες ανάγκες ουσιαστικά δικαιολογούν και έρχονται σε επίρρωση της ευρωπαϊκής πολιτικής για την αντιμετώπιση των κρίσεων. Όπου και πήγα στους τελευταίους έξι μήνες, στην Ινδία, στην Ταϊλάνδη, όπου είχε Βερμανούς ε, πρόσφυγες, στην Ιεμένη, στα σύνορα Τινησίας με Λιβύη, στα κατεχόμενα από το Ισραήλ ε, της Παλαιστίνης η ευρωπαϊκή ανθρωπιστική βοήθεια κάνει πράγματι τη διαφορά για χιλιάδες χιλιάδων ανθρώπων που γνωρίζουν ότι η Ευρώπη είναι μια δύναμη στον άξονα του καλού. Ότι εμείς τα πανούμε υπέρ των φτωχοτέρων και πιο ευθράφστων σημαντικά κονδύλια με στόχο να γίνει ο κόσμος μας ένα καλύτερο μέρος για όλους αλλά δεν πρέπει να δείξουμε χαλαρότητα, ιδίω σε στιγμές όπως η τωρινή. Και γι' αυτό το λόγο εγώ είμαι έτοιμη να προσαρμόσω και να αλλάξω τις πολιτικές μας για να ανταποκριθούν στις προκλήσεις που έχουμε ενώπιόν μας και στόχος μου σήμερα είναι να σας ενημερώσω σε σχέση με τις τέσσερις προτεραιότητες που σας παρουσίασα στην τελευταία μας συνάντηση ενίσχυσης ικανότητας αντιμετωπίσεως κρίσης, η αναθεώρηση του πλαισίου για τα ανθρωπιστικά θέματα, η δημιουργία ενός εθελοντικού <clears throat> ανθρωπιστικού σώματος στην Ευρωπαϊκή Ένωση και η πολιτική αρρωγής. Καταρχήν, διαχείριση καταστροφών. Η... Τα στοιχεία που έχουμε μας καταδεικνύουν πόσο σημαντική είναι η στάση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μια ιστοριούλα μονάχα που σας δείχνει τι έγινε. Η Ιαπωνία. Το Μάρτιο εγώ θα πήγαινα στην Ασία για να συμμετάσχω σε μία διεθνούς χαρακτήρα προσωμείωση για την απάντηση σε ένα σεισμό 7,5 ρίχτε που θα οδηγούσε ένα τσουνάμι που θα έπλητε την Ινδονησία. Ναι, πήγα στην Ασία αλλά έτυχε να βρεθώ ακριβώς στην Ιαπωνία όπως ο σεισμός του 9,0 δημιούργησε ένα ιδιαίτερα ισχυρό τσουνάμι και ένα πυρηνικό ατύχημα. Και κατάλαβα ότι η πραγματικότητα ήταν 100 φορές χειρότερη από την χειρότερη μας προσωμείωση. Γι' αυτό το λόγο θεωρώ ότι θα πρέπει να επιταχύνουμε την εφαρμογή της ανακοίνωσης για την απάντηση σε καταστροφές που έτυχε ομόφωνη υποστήριξη από τα κράτη-μέλη μα. Αυτό είναι ο λόγο για τον οποίο εμεί μέχρι το τέλο του 2011 θα καταθέσουμε προτάσει για τη μετάρρυθμιση του νομικού πλαισίου για την πολιτική προστασία <clears throat> και για το εργαλείο χρηματοδότησης ώστε να ενισχυθεί η ικανότητα απάντηση τη Ευρωπαϊκή Ένωση στι καταστροφέ, φυσικέ καταστροφέ. Ξεκινήσαμε μια δημόσια διαβούλευση με όλου του κύριου εμπλεκομένους και σε μια πρόσθετη συζήτηση στα μέσα Ιουνίου θα συζητήσουμε τα θέματα του, της αξιολόγησης. Θέλω να τονίσω πόσο μας ε, ενδιαφέρει και πόσο εξέρουμε το έργο της Επιτροπής σας, ιδίως το σχέδιο γνωμοδότησή σας για το οποίο είναι η γνωμοδότησή σας για την έκθεση της κυρίας Γκαρντίν για τις φυσικές καταστροφές. Εγώ είμαι ιδιαίτερα ευγνώμων στο Κοινοβουλίο για την υποστήριξή σας. Έχετε παίξει ηγετικό ρόλο για τα θέματα αυτά στο παρελθόν και σίγουρα θα το πράξετε και στο μέλλον. Τονίζουμε την βελτίωση της αποτελεσματικότητας μιας νέας συλλογικής απάντησης ώστε να εξασφαλίσουμε ότι η σωστή μορφή βοήθειας πηγαίνει ακριβώς εκεί που πρέπει να πάει στον ελάχιστο δυνατό τρόπο. Στόχος μας είναι να βελτιώσουμε την αποτελεσματικότητα το να συγκεντρώνουμε τις προσπάθειές μας και να, τις, ε, να κατανέμουμε το βάρος της προσπάθειας μεταξύ μας είναι απόλυτα σωστό και λογικό. Και εφόσον βασιζόμαστε σε μια θελοντική διαδικασία θα πρέπει να δώσουμε κίνητρα στα κράτη-μέλη για να έχουν ομάδες διαχείρισης κρίσης εν επιφυλακή για να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα τα οποία μπορούν να ανακύψουν. Και πάλι θέλω να τονίσω ότι συνεχώς κατανοώ τη σημασία του να βελτιωθεί η ορατότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κάνουμε καταπληκτικά πράγματα, αλλά συνήθως ο κόσμος δεν ξέρει τα κάνουμε. Η ενίσχυση λοιπόν της απάντησης για τις ε, <clears throat> φυσικές καταστροφές θα πρέπει να συμβαδίζει με την πρόληψη και την ετοιμότητα. Θα πρέπει να έχουμε ευρωπαϊκή αλληλεγγύη σε στιγμές φυσικής καταστροφής με ταχαία εθνικά μέτρα για να περιορίσουμε και να μετριάσουμε τον αντίκτυπο τέτοιων καταστροφών. Εκεί πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να καταλήξουμε σε προσπάθειες να υπάρξουν νομοθετικά μέτρα για τον μετριασμό των καταστροφών ήδη από του χρόνου. Και θέλω να τονίσω ότι κάθε ευρώ το οποίο επενδύεται σε προληπτικές δράσεις μπορεί να εξοικονομήσει 7 ευρώ σε έργο ανοικοδόμησης. Πάμε τώρα στο δεύτερο θέμα. Το πλαίσιο της ανθρωπιστικής μας δράσης. Με την ανακοίνωση του Δεκεμβρίου 2010 ξεκινήσαμε την ενδιάμεση αναθεώρηση σε σχέση με το σχέδιο δράση Ευρωπαϊκή Συνένεση όπου Χάρη στην έκθεση πρωτοβουλία της κυρίας Στρίφλερ, το Κοινοβούλιο συνέβαλε τα μάλα. Υπάρχει γενική συμφωνία ότι οι αρχές και οι στόχοι που περιλαμβάνονται στη συνένεση αυτή παραμένουν επίκαιροι και σημαντικοί. Πρέπει να διατηρήσουμε την επικέντρωση της ανθρωπιστικής μας δράσεις στις ανθρωπιστικές αρχές χωριστά και χωρίς καμία σχέση με τους στόχους της εξωτερικής πολιτικής και την γενική ατσέντα για την διαχείριση <clears throat> σε επίπεδο ασφάλειας και άμυνας των κρίσεων. Τρεις τομείς νομίζω ότι αξίζουν περισσότερη προσοχή. Η αποτελεσματικότητα της βοήθειας, συνεκτικότητα και συνοχή της δράσης Ευρωπαϊκής Ένωσης στα ανθρωπιστικά, ενίσχυση της συμμετοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς το Διεθνές Σύστημα Αντιμετώπισης Κρίσεων. Να σταθώ τώρα σε αυτά τα τρία θέματα, εν συντομία. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι είναι πάρα πολύ σημαντική ανθρωπιστική βοήθεια και ειδικότερα όταν αυτή αυξάνεται και μειώνονται οι πόροι. Ο καλύτερος τρόπος να εξυπηρετήσουμε όσους ζητούν, ε, όσους έχουν την ανάγκη μας, είναι να αυξήσουμε την ετοιμότητα της ανταπόκρισής μας. Χρειαζόμαστε καλύτερο καταμερισμό ε, φόρτου, καλύτερο καταμερισμό εργασίας. Ε, δηλαδή, δεν χρειάζεται να ασχολούμαστε μόνο με τις κρίσεις ε, οι οποίες χρηματοδοτούνται ε, και να παραγνωρίζουμε εντελώ όλες τις υπόλοιπες ε, που τελικά παραμένουν ορφανές. Και θα ήθελα να δεσμευθούν τα κράτη-μέλη να συμμετέχουν περισσότερο στον καθορισμό των επόμενων βημάτων που πρέπει να κάνουμε η αναθεώρηση του κανονισμού για την ανθρωπιστική βοήθεια που προβλέπεται στο πρόγραμμα εργασίας ε, για το 2011 ε, οφείλεται στο γεγονός ότι έχουμε ένα κανονισμό ήδη από το 1986 που μας εξυπηρετεί ε, καλά, όμως έχουν υπάρξει πολύ σημαντικές εξελίξεις από τότε και ειδικότερα μιλάω για τη νομική βάση για την ανθρωπιστική βοήθεια και το άρθρο 214 της Συνθήκης της Λισαβόνας όπως επίσης και την ε, υιοθέτηση της Ευρωπαϊκής Συνένεσης. Πρέπει λοιπόν να κάνουμε έναν απολογισμό του τι σημαίνει αυτό για μας και να αξιολογήσουμε τους κινδύνους και τα ωφέλη της ε, ε, επιπλέον νομοθεσίας. Πρέπει η ανθρωπιστική βοήθεια να προοδεύει και όχι να επαναχωρεί Γι' αυτό ακριβώς πιστεύω ότι και θα ήθελα να τονίσω ενώπιόν σας ότι θα πρέπει τα μέτρα που θα λάβουμε να είναι πολύ προσεκτικά ε, όσον αφορά την, το σχετικό κανονισμό. Θα αρχίσουν διαβουλεύσεις ε, κατά τους επερχόμενους μήνες ε, με τους εταίρους μας, με τα κράτη-μέλη και βεβαίως και με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Θα εκπονήσουμε πλήρη μελέτη αξιολόγησης αντικτύπου για να καθοδογήσουμε τις εργασίες μας και αν το κάνουμε αυτό σωστά η προσδοκία μου είναι ότι ε, δεν θα έχουμε βέβαια την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής πριν από τις αρχές του ερχόμενου έτους και θα ήθελα να σας ζητήσω να μας δώσετε το χρόνο να ε, το κάνουμε αυτό σωστά. Αυτή η νομοθετική αναθεώρηση που αφορά ε, τους στόχους και τους τρόπους εφαρμογής ε, ε, του καθορισμού των πολιτική, του, του καθορισμού των πολιτικών προκύπτει από το δημοσιονομικό πακέτο το τρέχον και θα επανέλθω σε αυτό σε λιγάκι δεύτερος τομέας της ε, μεσοπρόθεσμης αναθεώρησης ε, είναι η συνοχή και η συνέπεια της ε, αλληλεπίδρασης ανθρωπιστικής βοήθειας με άλλες κοινοτικές πολιτικές. Σεβόμενοι τον ανθρωπιστικό μας ρόλο και την εντολή μας πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι είναι συνεπής η ανταπόκρισή μας σε ευρωπαϊκό επίπεδο και υπάρχει ένα συγκεκριμένο θέμα το οποίο εμένα με ενδιαφέρει πάρα πολύ, δηλαδή μεγαλύτερη σχέση και περισσότερη, περισσότερο περισσότερος δεσμός, μετα, περισσότερη σύνδεσμη μεταξύ της ανθρωπιστικής βοήθειας και της ανάπτυξης. Δηλαδή, οι άνθρωποι οι οποίοι ε, έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές, να έχουν κατεπίγουσα βοήθεια, η οποία ε, πηγαίνει ακριβώς σε επιχειρήσεις ανακούφισης αλλά και στην ανάπτυξη. Δηλαδή, σώζουμε ζωές, αλλά δεν αφήνουμε και τον κόσμο στη μοίρα του, δηλαδή ε, δεν τους αφήνουμε μετά στη μοίρα τους όταν πια δεν υπάρχει ανθρωπιστική βοήθεια. Προσπαθούμε να δούμε και τη μετέπειτα κατάσταση και πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να το κάνουμε αυτό καλύτερα. Μία ευκαιρία την οποία εντοπίσαμε είναι η ακτή ελεφαντοστού, δηλαδή προσπαθήσαμε να δείξουμε ότι έχουμε μία συνολική προσέγγιση για την ανακούφιση, την ανοικοδόμηση και την ανάπτυξη. Αποκινούμε τον Επίτροπο Τίμπαλξ. Ε, αναγνωρίσαμε ότι αυτή η ομάδα ε, της ε, ανακούφισης, της αποκατάστασης και της ανάπτυξης ε, λειτουργεί μεν καλά, αλλά πρέπει να υπάρχει ένα πλαίσιο πολιτικής που δίνει μεγαλύτερη δυνατότητα ευελιξίας των πολιτικών σε ένα μεταβατικό πλαίσιο. Και το τρίτο που θα ήθελα να θέσω είναι η ενισχυμένη συνεισφορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Διεθνές Ανθρωπιστικό Σύστημα. Είμαστε πραγματικά ο πρώτος ανθρωπιστικός δωρητής και έχουμε την υποχρέωση να χρησιμοποιήσουμε όλο μας το βάρος για να επηρεάσουμε τη διεθνή ανθρωπιστική ατζέντα. Καταλαβαίνω ότι έγινε και μία ε, παρουσίαση από τον Άντριου Μίτσελ εχθές ε, σε σχέση με την επισκόπηση ε, της ανθρωπιστικής βοήθειας και συμφωνώ απόλυτα με το στόχο που προέκυψε από την αναθεώρηση αυτή. Χρειαζόμαστε καλύτερη αποδοτικότητα, εναρμόνιση των στόχων, καλύτερη συνεργασία και η άποψή μου είναι ότι πρέπει να υπάρξει μια διαδικασία με διεθνή συνένεση ισχυρή που μπορεί να είναι παρόμοια με αυτή των αναπτυξιακών στόχων της χιλετίας προκειμένου να καθοδηγήσουμε τις εργασίες μας. Θα με ενδιαφέρε πάρα πολύ να, μας, να, να ακούσω και τη δική σας άποψη σε σχέση με το θέμα αυτό. Έχουμε μια πραγματική ευκαιρία του χρόνου. Θα έχουν περάσει 20 χρόνια από τότε που υπάρχει το ΕΚΟ, το Ανθρωπιστικό Γραφείο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και μπορούμε αυτήν την 20η επέτειο να τη χρησιμοποιήσουμε όχι μόνο για να προβληματιστούμε για το παρελθόν, αλλά πολύ περισσότερο για το μέλλον. Να δούμε δηλαδή πώς μπορούμε να ενισχύσουμε την ανθρωπιστική μας ατζέντα. Μία βασική προτεραιότητά μου είναι το εθελοντικό ανθρωπιστικό σώμα η Ευρωπαϊκή Ένωση το εθελοντικό αυτό σώμα είναι μια πολύ μεγάλη ε, δέσμευση ε, γιατί είναι πολύ, ε, είναι πολλοί εθελοντές που ε, εμπλέκονται και βλέπω ότι πάρα πολλοί κόσμος θέλει πράγματι εθελοντικά να βοηθήσει τους συνανθρώπους του. Ε, είχαμε και μια ανακοίνωση το 2010 βάσει της οποίας είχαμε αποφασίσει να ξεκινήσουμε με μια πιλωτική φάση που θα μας έδινε τη δυνατότητα το 2011 να καταλήξουμε σε ένα πραγματικό σώμα ανθρωπιστικής δράσης, επιλογή των εθελοντών, ε, εκπαίδευση και ανάπτυξη του. Μέχρι το τέλος του Ιουνίου θα έχουμε πλήρως οργανωμένη και ε, θα λειτουργεί πλέον αυτή η πρώτη πιλωτική φάση και επί τη βάση της πιλωτικής αυτής εμπειρίας θα παρουσιάσουμε την νομοθετική πρωτοβουλία μας ε, το 2012. Τελευταία και τέταρτη και τελευταία προτεραιότητα η οποία είναι εξίσου σημαντική είναι η ενίσχυση της επιζητιστικής ε, βοήθειας και η σχετική μας πολιτική είναι γεγονός ε, ότι έχουμε αφήσει πίσω μας τις δεκαετίες ε, ε, κατά τις οποίες είχαν μειωθεί οι τιμές των τροφίμων. Τώρα αυτή τη στιγμή έχουμε περάσει σε μια φάση ανωδικής τάσης της τιμής των τροφίμων με την κλιματική αλλαγή και με την πίεση της ανάπτυξης της μεσαίας τάξης στον αναπτυσσόμενο κόσμο, δεν υπάρχει κανένας λόγος να θεωρούμε ότι μπορούμε να αποφύγουμε αυτήν την ενωδική τάση και γι' αυτό ακριβώς η ασφάλεια η διατροφική είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό ζήτημα για πολύ κόσμο. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν ε, συμμετείχαμε πάρα πολύ στον εξυγχρονισμό της ε, επαναδια... της Σύμβασης του 1999 για την επιστημιστική βοήθεια βλέπω ότι θα το συζητήσετε και σήμερα. Είμαστε πραγματικά πρωτοστάτες στη συζήτηση αυτή. Έχουμε κάνει πολύ σημαντική πρόοδο για το βασικό ζήτημα της Σύμβασης που είναι ουσιαστικά η επιστημιστική βοήθεια να καταστεί ένα ε, μέσο ελεύθερο από το τοπικό lobbying και από τις πιέσεις του τοπικού lobbying. Έχουμε δηλαδή πάρει την απόφαση ότι δεν θα, δεν θα πιέσουμε τα γεωργικά μας πλεονάσματα ως επιστηστική βοήθεια. Ε, πρέπει να πω ότι ο Καναδάς ε, συμφωνεί με την άποψή μας και οι Ηνωμένε Πολιτείε που ήταν πολύ πιο δύσκολο να πιστεί επιτέλους μετακινήθηκε από τη θέση της και έχει κάνει πολύ σημαντικά βήματα προς τη δική μας άποψη. Ένα πολύ σημαντικό ζήτημα λοιπόν είναι το ζήτημα της διατροφής και επ' αυτού του ζητήματος ε, θέλουμε να προωθήσουμε την, ε, το πρόγραμμα των πολιτικών, των πολιτικών μας. Θα ήθελα να ευχαριστήσω το Κοινοβούλιο γιατί ενδιαφέρεται πολύ για αυτό το θέμα της ε, ε, επισητιστικής βοήθειας και θα ήθελα να ευχαριστήσω και τους συναδέλφους της, ε, από την πλευρά της ανάπτυξης που ασχολήθηκαν με αυτό το θέμα. Για παράδειγμα, η εργασία της Γκαμπριέλ Τσίμερ είναι πάρα πολύ σημαντική για το θέμα αυτό της επισητιστικής βοήθειας. Και ολοκληρώνοντας θα ήθελα να πω ότι σήμερα έχουμε και τη συζήτηση για το ε, πολιετές ε, ε, πρόγραμμα. Εμείς θα υποβάλουμε τις προτάσεις μας μέχρι τα τέλη του Ιουνίου για, το, για τις διοργανικές διαπραγματεύσεις και προκειμένου να ξεκινήσουν αυτές. Τώρα, ποιος είναι ο δικός μου ρόλος για αυτές τις τέσσερις προτεραιότητες. Έχουμε να αντιμετωπίσουμε πολύ σοβαρές πιέσεις ε, στην χρηματοδότηση των εργασιών μας. Ο τρέχον προϋπολογισμός μας προφανώς δεν επαρκεί και το βλέπετε ε, χρόνο με το χρόνο. Κάθε φορά πρέπει να αντλήσουμε από το αποθεματικό περισσότερα χρήματα. Εγώ προέρχομαι από εγώ είμαι υπέρμαχος μιας ε, ε, υπεύθυνης δημοσιονομικής ε, φιλοσοφίας, για να το πω έτσι, και πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί, ειδικότερα όταν υπάρχουν άνθρωποι που υποφέρουν στις χώρες τους. Η δική μου έκκληση θα ήταν να προσεγγίσουμε ως εξής τον προπολογισμό μας, να εξασφαλίσουμε ότι αντικειμενικά παρέχουμε χρηματοδότηση η οποία ε, είναι σε αναλογία με τις ε, ιστορικές μας παραδόσεις και τις ανάγκες ε, των, του, του πληθυσμού, περίπου ένα δισεκατομμύριο κατέτος και επίσης να εξασφαλίσουμε ότι έχουμε μια πολύ προσεκτική γραμμή αποθεματικού, κάθε φορά δηλαδή που υπερβαίνουμε πολύ ε, τις ε, δυνατότητές μας. Και αυτό έχει συμβεί 9 στις 10 φορές τα τελευταία 10 χρόνια. σε όσες χώρες και αν έχω πάει, ε, εντός, εκτός ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης, ε, πάντοτε ήταν σαφές για μένα ότι η Ευρώπη έχει κερδίσει το σεβασμό των πολιτών μας, 80% είναι υπέρ της δουλειάς μας και μιλάω για τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν πληγεί από διάφορες καταστροφές σε όλο τον κόσμο. Αυτό γιατί ακριβώς βασιζόμαστε στην αρχή στην αξία της αλληλεγγύης, γιατί πιστεύουμε ότι αυτό είναι το σωστό. Αυτό πρέπει να κάνουμε. Όμως γίνεται πιο περίπλοκος και πιο ε, εύθραυτος ο κόσμος μας και γι' αυτό είναι και το σωστό ε, να ε, η ανθρωπιστική βοήθεια είναι κάτι σωστό για τη σταθερότητα των κοινωνιών σε οποίες διαβιούν οι πολίτες μας. Ευχαριστούμε. Να δώσω το λόγο στους συναδέλφους. Δίνω το λόγο στον εαυτό μου λοιπόν. Θα, μου, θα με παρακαλέσω να είμαι σύντομη. Κυρία Επίτροπε, με προλάβατε σε κάποια από τα ερωτήματα που σκόπευα να σας θέσω. Όταν προτείνεται αναθεώρηση του κανονισμού για την ανθρωπιστική βοήθεια που χρονολογείται από το 1996, η αναθεώρηση αυτή πρέπει να γίνει και σε σχέση με την ευρωπαϊκή συμφωνία για την ανθρωπιστική βοήθεια εφόσον υπάρχει. Πιστεύετε ότι κάποια κράτη-μέλη μπορεί να επαναχωρήσουν σε σχέση με κάποιου από του στόχου και τα σχέδιά μας επίσης διασύνδεση της επίγουσας βοήθειας και το οικοδότησής μας με μέσα, διότι υπάρχει εδώ επικάλυψη των πολιτικών προσπαθειών. Πώς θα διαμορφωθεί η προσπάθεια για την ευελιξία και την συμπληρωματικότητα των δημοσιονομικών μέσων που υπάρχουν, καθώς και τη μεταβατική φάση μεταξύ κατεπίγουσας ανάγκης και ανάπτυξης. Πώς έχει προχωρήσει η μελέτη στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής εν ώψη και των ερχόμενων δημοσιονομικών προοπτικών και της αναθεώρησης του κανονισμού για την ανθρωπιστική βοήθεια. Και ολοκληρώνω οργανώσατε πρώτο γύρο διαβουλεύσεων με τους ε, ενδιαφερομένους για την προετοιμασία νομοθετικών προτάσεων που θα αναθεωρήσουν τα μέτρα πολιτικής προστασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και φάνηκε ότι τα κράτη-μέλη είναι μάλλον υπέρ της δημιουργίας ενός ε, κέντρου αντίδρασης της Ευρωπαϊκής Ένωσης που να βασίζεται στις δυνατότητες των κρατών μελών και εθελοντικά να συμμετέχει στις δράσεις της Ένωσης. Το ερώτημά μου λοιπόν είναι πώς ε, θα διασφαλίσετε αυτήν την εθελοντική διάθεση των μέσων του κέντρου. Κάποια κάτι μέλη τάχθηκαν υπέρ ελκυστικών μέτρων, όπως για παράδειγμα αυτόματες η χρηματοδότηση των μεταφορικών μέσων κτλ. κτλ. Να περάσω σε μια άλλη ερώτηση. Να ακούσουμε πρώτα δύο-τρεις συναδέλφους, κυρία Κρατσού. Ευχαριστώ. Κατά πρώτον να σας ευχαριστήσω κυρία Επίτροπε που είστε εδώ. Ξέρετε ότι είναι πολύ σημαντικό για μας να έχουμε αυτό το διάλογο και αυτή τη συνοπτική εικόνα της όλης κατάστασης. Σας ευχαριστούμε λοιπόν για το πόσο πρόθυμα έρχεστε κοντά μας. Πάντως τα μέλη της Επιτροπής Ανάπτυξης και κυρίως εγώ η ίδια πρέπει να τονίσω την πρότασή μας για την ανθρωπιστική βοήθεια για το 12. Όπως είπατε και εσείς, υπάρχουν πολλές καλές ιδέες. Θα θέλαμε λοιπόν ο διάλογος να διευρυνθεί. Και η ανακοίνωση του 2010 για την ισχυρότερη ευρωπαϊκή απόκριση στις ε, ε, κρίσεις για την ανθρωπιστική βοήθεια και την αντιμετώπιση τους να ανανεωθεί θέλουμε το κέντρο για την πολιτική προστασία να δημιουργηθεί, να ενισχυθούν οι υπάρχοντες μηχανισμοί και να υπάρξουν διευθετήσεις για την συνεργασία μεταξύ της, Επιτροπής, της Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της ίδιας της Επιτροπής. Χρειάζεται εδώ συνένεση η οποία μπορεί να μας ε, έρχεται και από την απόφαση του 2007 για την ανθρωπιστική βοήθεια. Και εδώ βεβαίω μπορούμε να υπολογίζουμε και στη βοήθεια τη Υπηρεσία Εξωτερική Δράση και χάρη στου θεωρητικού και του διπλωμάτε των ευρωπαϊκών κρατών. Χρειάζεται εδώ μια ευρωπαϊκή προσέγγιση στην ανθρωπιστική βοήθεια. Θέλουμε και αναθεώρηση του κανονισμού για την ανθρωπιστική βοήθεια τη Ευρωπαϊκή Ένωση, κάτι που προβλέπει για το τελευταίο τρίμηνο του 2011 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Επίσης θα πρέπει να υπάρξουν μέτρα ε, ως κατεξουσιοδότηση πράξης ε, για να ενισχυθούν τα δημοσιονομικά μέσα και οι ανθρωπιστικές δράσεις που ως τώρα δεν ε, χρηματοδοτούνται επαρκώς. Είδαμε ότι μέσα στα έτη και στα χρόνια με το πέρασμα των καιρού δεν αρκεί ετησίως η πρικοδότηση που έχουμε προβλέψει. Πρέπει να έχουμε αυστηρός ανθρωπιστικούς στόχους και να ασχοληθούμε με την πρόληψη των φυσικών καταστροφών, τις καταστάσεις, ε, τις περιπτώσεις μετάβασης και την ανακούφιση από κρίσεις ή την προσπάθεια αναχέτησης και μείωσης των φυσικών καταστροφών. Θα πρέπει η μείωση αυτή στις αναπτυσσόμενες χώρες να επιδιωχθεί με μια σχετική, ένα σχετικό κατάλογο προτεραιοτήτων της αναχέτησης των καταστροφών. Θα μεταφέρουμε και γενικότερα τις προτάσεις της ομάδας μας, αλλά ελπίζω με το πρόγραμμά σας και με τη γραμματεία να λάβουμε υπόψη το κατά πόσον ε, τα κράτη-μέλη εκπληρώνουν τις υποχρέσεις τους ως προς την ανθρωπιστική βοήθεια. Για την ώρα μόνο εκεί προς τα καταφέρνει αυτό. Είναι θέμα κουλτούρας και πολιτιστικής ε, καινοτροπίας της χώρας μας. Θα πρέπει λοιπόν να το επιδιώξουμε. Θα έπρεπε να οργανωθεί μια διμερίδα του χρόνου συναντήσεις, συζητήσεις, όχι μόνο με κυβερνήσεις, αλλά και με κυβερνητικές οργανώσεις από τα νέα κράτη-μέλη για να κινητοποιηθούν. Ελπίζω ότι οι συνάδελφοί σας θα... και οι συνάδελφοι εδώ θα καταλάβουν την ανάγκη και οι χώρες αυτές να κρατούν τις υποσχέσεις τους. στις ε, βόρειες χώρες της Ευρώπης, στις σκανδιναβικές, υπάρχει λόγω χάρη τελείως διαφορετική φιλοσοφία από τη στη δική μας. Ευχαριστούμε κυρία Κρετσού, ο κυρία Κέλλερ. Ευχαριστούμε. Η Κύπρος μπορεί να μειώνει πολύ και το κόστος της ε, αναπτυξιακής βοήθειας εφόσον τα μετρήσει κανείς βέβαια και με διαφορετική μέθοδο. Ευχαριστούμε λοιπόν κυρία Ντόρτιβα εδώ για την παρουσίαση του προγράμματος εργασιών σας. Για το θέμα της πρόληψης όμως ε, καταστροφών, το θέμα είναι τι θα γίνει μετά την πρώτη λόγου χάρη παροχή βοήθειας, το πρώτο κονδύλι. Ίσως πρέπει να υπάρχει κάποια είδους ενημέρωση, κάποια αναγγελία, να ξέρουμε και τι αποτελέσματα υπήρχαν από τις συζητήσεις. Δεν θα έπρεπε να υπάρχει συμμετοχή και επίσημη. Έπειτα, διερωτώ με κατά πόσον από πέρσι που είχαμε πολλέ τέτοιε καταστροφέ και είχατε κι εσεί πολλή δουλειά. Αντλήσατε διδάγματα από όλε αυτέ τι εμπειρίε. Ίσως σε κάποιε περιπτώσει να είπατε, να, αυτό θα έπρεπε να έχει γίνει διαφορετικά ή να γίνει διαφορετικά στο μέλλον. Κάτι τέτοιο. Και επίση συζητήσαμε για την περίπτωση τη Λιβύη, όπου και πάλι προέκυψε το θέμα. Ανθρωπιστική βοήθεια μεν, αλλά με στατιστική προστασία ε, ταυτόχρονα. Τι άποψη έχετε εδώ. Συμφωνείτε με μια τέτοια είδου πρόταση. Τέλος, επειδή αναφέρατε και την αποτελεσματικότητα και την ε, επικείμενη συνάντηση στην, ε, στην Βουσά. Τι πιστεύετε ότι θα πρέπει να συζητηθεί από την άποψη της ανθρωπιστικής βοήθειας και της ανθρωπιστικής βοήθειας. Ο κύριος Σφένσον. Thank Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε πάντα μας ενθαρρύνει και μας εντυπωσιάζει η συνάντηση και το άκουσμα της κυρίας Επιτρόπου. Σας ευχαριστώ που ήρθατε και επικροτώ και το μήνυμα της ε, αλληλεγγύης όπου τα είπατε ότι πρέπει να κοιτάμε προς, τα, προς το μέλλον όχι προς το παρελθόν. Συμφωνώ με αυτά που είπατε για το συντονισμό και την ανάγκη να έχουμε μια πιο μακροχρόνια σχεδίαση. Θα ήθελα τώρα να σας ρωτήσω τα εξής κυρία Επίτροπε, αν θέλετε να μας δώσετε πιο πολλές λεπτομέρειες για τα συγκεκριμένα σχέδια για το συντονισμό και την ευκαμψία της βοήθειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να μειώσουμε το χάσμα το οποίο υπάρχει μεταξύ της, της ε, ανθρωπιστικής και της ε, αναπτυξιακής βοήθειας και να μειωθούν και τα ε, αποτελέσματα αυτού του χάσματος. Κύριε Τσόζεβα, σας προτείνω να λάβετε το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ για τα ερωτήματά σας και τα σχόλιά σας. Σε αυτά που είπε η κυρία Στίφλερ. Έχουμε ένα κανονισμό το κανονισμό του 1996 που έχει λειτουργήσει καλά και εξακολουθεί να λειτουργεί θετικά. Έχουμε κάνει ένα απολογισμό, έχουμε κάνει μια εξέταση εφαρμογή αυτού του κανονισμού και έχουμε διαπιστώσει ότι σε σχέση με τους κύριους στόχους και την επίτευξή τους είναι καλός κανονισμός. Προφανώς θα μπορούσαμε να προχωρήσουμε περισσότερο μετά και από τις θεσμικές αλλαγές που έχουν γίνει, μετά από την αλλαγή του πρώτου εργασίας μας, με την ανάδυση νέων χορηγών και νέων αναγκών. Όλα αυτά πρέπει να τα κάνουμε όμως με κάποια σοφροσύνη. Γιατί όταν ξεκινήσουμε κάτι τελείως καινούριο, όταν ανοίξουμε τους ασκούς του αιώλου, μπορεί να προέλθουν και αλλαγές οι οποίες δεν είναι αυτές που επιζητούμε και δεν είναι αυτές που είναι επικοδομητικές και μας βοηθούν για το μέλλον. Αυτό που βλέπουμε αυτή τη στιγμή σε πολλά κράτη-μέλη για, για μια πολυπικιλία λόγων. Είναι ένα κίνδυνος για τα πιο κρίσιμα στοιχεία της ανθρωπιστικής μας προσέγγισης που είναι μια προσέγγιση βάση αναγκών. Γιατί πρέπει να ακολουθήσουμε μια τέτοια προσέγγιση. Για μας είναι προφανές, αλλά κάποιοι άλλοι μερικές φορές μπορεί να μην καταλαβαίνουν τι σημαίνει κάτι τέτοιο. Η προσέγγιση βάση αναγκών σημαίνει ότι δεν κοιτάμε τη θρησκεία, δεν κοιτάμε τις πολιτικές πεπιθήσεις. Το μόνο πράγμα το οποίο κατευθύνει τη δράση μας είναι τα βάσανα των ανθρώπων, τα οποία προσπαθούμε εμείς να ανακουφίσουμε. Με αυτόν τον τρόπο, εμείς οι Ευρωπαίοι, ακολουθώντας μια τέτοια προσέγγιση, επιτυχάνουμε δύο σημαντικούς στόχους. Καταρχήν φυσικά να βοηθήσουμε αυτούς οι οποίοι χρειάζονται βοήθεια και έτσι ενισχύουμε και τη σταθερότητα και την ειρήνη στον κόσμο, αλλά κατά δεύτερο λόγο δίνουμε ένα παράδειγμα και για τους άλλους. Αυτό είναι η ανθρωπιστική βοήθεια τους δείχνουμε. Δεν είναι πολιτικό εργαλείο. Δεν είναι ένα σύστημα μέσω του οποίου προσπαθούμε να επιβάλλουμε τις πολιτικές μας ή τις σκεφτικές πεπιθήσεις. Όχι, είναι ένα εργαλείο για να βοηθήσουμε τα άτομα που δοκιμάζονται. Αυτή είναι μια αρχή λοιπόν την οποία εμεί θα πρέπει να την προασπίσουμε. Εγώ ένιωσα να με ενθαρρύνει πάρα πολύ το γεγονός ότι πριν από λίγες μέρες ήμουνα στη Ρωσία, με συναντήθηκα με τον κύριο Σόιγκουν, τον Υπουργό για έκτακτη, αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και τον Υπουργό Εξωτερικών της Ρωσίας και μας είπαν ότι οι Ρώσοι θέλουν να μην είναι πολιτικού χαρακτήρα η ανθρωπιστική <clears throat> βοήθεια. Είναι λοιπόν σύμμαχοί μας γιατί έχουν και αυτοί μια αρνητική εμπειρία από το παρελθόν για τα θέματα αυτά. Αν ρωτάτε ποιοι είναι οι κίνδυνοι. Για μένα αυτό είναι ο πιο μεγάλο κίνδυνος. Πολιτικοποίηση τη βοήθεια. Μπορεί να έχουν την εντύπωση ότι είναι καλύτερα να τα βάλουμε όλα μαζί. Εξωτερική πολιτική, ε, εμπορική πολιτική, αναπτυξιακή πολιτική, ανθρωπιστική βοήθεια. Το λένε αυτό καλή την πίστη. Αλλά ξέρουμε ότι πολλές φορές ότι ο δρόμος για την κόλαση έχει στρωθεί με καλές προθέσεις. Είναι ένα με καλών προθέσεων. Λοιπόν, εμείς θέλουμε να εξετάσουμε και πάλι αυτόν τον κανονισμό, αλλά με ένα σαφές σχέδιο, μια σαφή στρατηγική για το πώς θα πρέπει να γίνει αυτή η αναθεώρηση. Και εδώ είναι πολύ σημαντικό να σκεφτούμε το τι θα γίνει το 2012 και όχι μονάχα μέχρι το τέλος του 2011 δεν θέλουμε να βάλουμε τον εαυτό μας σε χρονική πίεση, μπορεί να μας εμποδίσει να κάνουμε τις κατάλληλες αλλαγές για την ευκαμψία και τη συμπληρωματικότητα των εργαλείων που υπάρχουν ήδη. Προφανώς προσπαθούμε να εξασφαλίσουμε ανεξαρτησία και ουδετερότητα, αλλά αυτό σαν τμήμα μια γενικής εμπλοκής Ευρωπαϊκής Ένωσης σε πολύπλοκες καταστάσεις. Η συμπληρωματικότητα αφορά κυρίως τα εργαλεία ανάπτυξης, τα εργαλεία σταθερότητος και στο πλαίσιο αυτό, αυτό που διαπιστώνουμε είναι ότι τα εργαλεία σταθερότητα είναι <clears throat> εύκαμπτα. Μπορούμε να συνδυάσουμε πολύ εύκολα αυτά που κάνουμε με αυτά τα οποία κάνουν τα εργαλεία σταθερότητα. Αλλά αυτό δεν αφορά ένα μεγάλο κομμάτι της αναπτυξιακής βοήθειας που χρειάζεται μακρό χρόνο προετοιμασίας, μακρό χρόνο εφαρμογής και πέφτουμε στο κενό αυτό, στο χάσμα που αναφέρατε εδώ. Σε ένα ιδανικό κόσμο θα έπρεπε να υπάρχει κάποιος ενδιάμεσος χώρος, όχι κατά να ένα νέο εργαλείο, από ό,τι καταλαβαίνω τα τωρινά μας εργαλεία αν θέλαμε θα μας επέτρεπαν να διευρύνουμε τον χώρο χρηματοδότησης για να υπάρχει μεγαλύτερη ευκαμψία στη χρηματοδότηση των μέτρων μας. Και νομίζω ότι είναι το ερώτημα που έθεσε ο κ. Σουάνης και η κυρία Κρετούντ για το πώς μπορούμε να βελτιώσουμε τα πράγματα στον τομέα αυτό. Τα δικά μου συμπεράσματα είναι πρώτα απ' όλα θα πρέπει να, να δημιουργήσουμε ένα δημοσιονομικό χώρο στα πλαίσια της ανάπτυξης, δηλαδή να έρχεται με μεγαλύτερη ευκαμψία και ταχύτερα χρηματοδότηση. Δεύτερον, θα πρέπει να δώσουμε κίνητρα και πιέσεις ώστε να υπάρχει και ανθρωπιστική βοήθεια και σε αναπτυξιακό επίπεδο βοήθειας και να υπάρξει συνεργασία των εμπειρογνωμόνων και από τις δύο πλευρές. Έχουμε εργαλεία λοιπόν για αντιμετώπιση καταστροφών που συναθρίζουν όλους τους εμπλεκομένους, φτάνουμε σε κάποιο σημείο στην σχεδίαση, αλλά μετά θα πρέπει να αφασίσουμε και πώς θα γίνει η εφαρμογή των σχεδίων. Και αυτά ισχύουν και για τις δύο πλευρές. Εγώ έχω έρθει από την πλευρά της ανάπτυξης, τώρα είμαι στην ανθρωπιστική πλευρά. Οι εργαζόμενοι στον αναπτυξιακό τομέα θεωρούν ότι είναι απλώς πυροσβέστες αυτοί που εργάζονται στον ανθρωπιστικό τομέα, αλλά δεν καταλαβαίνουν το πώς θα εξαλειφθούν οι ρίζες της ε, ένδυας και αυτοί που εργάζονται στον ανθρωπιστικό τομέα θεωρούν ότι αυτοί που δουλεύουν στην ανάπτυξη βραδιπορούν και αργούν πάρα πολύ. Και εγώ είχα πει στον κύριο Σέλικ, το πρώην αφεντικό μου, ότι θα πρέπει για τι παγκοσμίε, Τράπεζε, ότι πρέπει να ενθαρρύνουμε μια ευκαμψία σε δύσκολε καταστάσει. Να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε καταστάσει μετά από μια κρίση, μετά από μια καταστροφή, να φέρουμε τις δύο κοινότητες, τους ανθρωπιστές και τους αναπτυξιστές, στο σωστό επίπεδο, ώστε να υπάρξει μια κοινή ηγεσία και από τις δύο πλευράς και αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό στην περίπτωση των λεγόμενων ευθραύστων κρατών. Και τρίτο σημείο, θα πρέπει να έχουμε ένα βαθμό λογικό πίνακα που να λέει «Να, εδώ έχουμε την κατάσταση ενός κράτους που είναι σε εύθραυστη κατάσταση και να μπορούμε να κρίνουμε από τη βάση των ενεργειών μας τι προκύπτει». Και επίσης για τους πολίτες, για τους φορολογούμενους της, Ευρώπης. Εγώ έχω αναλάβει την ευθύνη ότι όλα αυτά τα οποία δαπανούνται στον ανθρωπιστικό τομέα έχουν σαν πρώτη, στο μέρη, πρώτη στη μέρημνα το να σώσουμε ζωές, όχι για να εκπαιδεύουμε τα παιδιά. Σε τρία χρόνια θα έρθει κάποιος από το γραφείο του κυρίου Πίμπολ να ζητήσει να υπάρξει ένα σχέδιο εκπαίδευσης. Μα δεν μπορούμε να δουλεύουμε έτσι. Λοιπόν, Συνοψίζοντας, πρέπει να σχεδιάζουμε από κοινού, πρέπει να συνεννοούνται οι, οι δικοί μας, να εκπαιδεύονται μαζί, να υπάρχει λογοδοσία σε σχέση με τα αποτελέσματα, να ξέρουμε τι θα κάνουμε. Για την ακτή του αλεφαντοστού έχουμε περίπου 60 εκατομμύρια από ε, την πλευρά την ανθρωπιστική, 180 από την ανάπτυξη και αυτό σημαίνει ότι πρέπει να χρησιμοποιήσουμε αυτά τα χρήματα για να δοθούν θέσεις εργασίας. Να μπορούν να τρώνε οι άνθρωποι. Για να τρώνε χρειάζονται λεφτά. Δεν πρέπει να τους δώσουμε τα λεφτά για να τρώνε, πρέπει να τους δώσουμε λεφτά ώστε να εργάζονται μέσω θέσεων εργασίας και έτσι να εξυπηρετήσουμε στόχους αναπτυξιακούς. Αυτοί είναι οι τρόποι με τους οποίους εμείς μπορούμε να πετύχουμε πρόοδο στον τομέα αυτό. Για τις νομοθετικές προτάσεις για την ενίσχυση της ε, ικανότητας αντιμετώπισης κρίσεων. Αυτό το οποίο θέλουμε να κάνουμε είναι να περπατάμε και με τα δύο πόδια, λέει η κυρία Επίτροπος. Καταρχήν να δούμε για πράγματα που δεν χρειάζονται νομοθετικές ρυθμίσεις, όπως το να έχουμε ένα Ευρωπαϊκό Κέντρο Άμεσης Αντιμετώπισης Κρίσεων, που να χρησιμοποιήσει τις ομάδες μας για ανθρωπιστική ανακούφιση. Αυτό ζητάει ένα νομοθετικό πλαίσιο, αλλά είναι μια πλατφόρμα που μπορεί να μας βοηθήσει να ολοκληρώσουμε καλύτερα τη χρήση των εμπειρογνωμών από τα κράτη-μέλη. Αλλά χρειαζόμαστε μια νομοθετική πρόταση. Όταν έρθουμε να σας θα πούμε να τι έχουμε από τις υποσχέσεις των κρατών μελών για να δημιουργηθεί αυτή η δύναμη, εδώ είναι τα κενά και έτσι προτείνουμε να γεμίσουμε και κενά τα οποία υπάρχουν. Και ίσως θα μπορούσαμε να έχουμε περισσότερα κίνητρα προς τα κρατημέλη να τους δίδουμε κάποιο, κάποια απόδοση κόστους για τις μεταφορές του προσωπικού ή με το να έχουμε κάποιες άλλες πτυχές οι οποίες τους ε, ενισχύουν το έργο τους. Δεν ξέρω λοιπόν συνολικά πώς θα είναι. Αλλά όταν έρθουμε ενώπιον του Κοινοβουλίου θα είναι πολύ σημαντικό να έχουμε την υποστήριξή σας. Είσαστε τμήμα της διαδικασίας σχεδιασμού ώστε να δημιουργηθεί ένα σύστημα το οποίο λειτουργεί. Όπως μας είπανε οι 93% των ανθρώπων που συναντήσαμε θέλουν όλη η Ευρώπη να λειτουργεί από κοινού για να αντιμετωπίσει τις καταστροφές. για αυτά που είπε η κυρία για την κατανομή αρμοδιοτήτων με την υπηρεσία εξωτερικών θεμάτων. Εμείς είμαστε οι πρώτοι οι οποίοι ανταποκρινόμαστε σε μια έκτακτη κατάσταση. Εμείς είμαστε οι πρώτοι που πηγαίνουμε στον χώρο της καταστροφής. Δίνουμε ανθρωπιστική ανακούφιση. Εξασφαλίζουμε την πολιτική προστασία ή δυνατόν θεσπίζουμε ένα μηχανισμό συντονισμού για τα κρατη ώστε να μπορούν να αναπτύξουν τις ε, ομάδες αντιμετώπισης. Και αν τώρα είναι μια καταστροφή εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχουμε σύνδεση με την υπηρεσία εξωτερικής δράσης, αν υπάρχει πολιτική διάσταση ή διάσταση άμυνας, τότε είναι δικός τους ρόλος. Τόσες φορές το έχουμε κάνει, που νομίζω ότι ξέρουμε καλά ποιος είναι ο ρόλος μας και πώς θα πρέπει να τον διαδραματίσουμε. Με ρωτήσατε σήμερα το πρωί στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων κάτι που μπορεί να σας ενδιαφέρει. Το ερώτημα είναι, πρέπει να υπάρχει μονάχα ένα κέντρο για αντιμετώπιση κρίσης. Να υπάρχει ένα κέντρο το οποίο αντιμετωπίζει όλες τις κρίσεις, είτε είναι πολιτικές, είτε είναι αμυντικούς, αμυντικού χαρακτήρα κτλ. Και από αυτά τα οποία έχουμε δει στα κράτη-μέλη ή σε άλλα, άλλες, άλλα κράτη όπως οι ΗΠΑ και η Ρωσία, η απάντησή μου είναι όχι. Θέλουμε ένα σύστημα για τα ανθρωπιστικά και την πολιτική προστασία που να ασχολείται μόνο με τα θέματα αυτά. Γιατί αυτοί που ασχολούνται με τα θέματα αυτά είναι αυτοί που πρέπει πρώτα απ' όλους να δώσουν μια απάντηση σε μια κρίση. Και πρέπει από την άλλη μεριά να έχουμε ένα πολιτικό στρατιωτικό κέντρο αντιμετώπισης κρίσεων στο οποίο θα πρέπει και εμείς να έχουμε κάποια συνεισφορά. Να μπορώ εγώ να είμαι μέλος αυτού του Συμβουλίου όταν πρέπει να αποφασίσει για στρατιωτική αντιμετώπιση. Και αν θυμόσαστε όταν ο πρόεδρος Ομπάμα παρακολουθούσε τις επιχειρήσεις κατά του Μπιν Λάντεν το έκανε στο Λευκό Οίκο αλλά μπορεί να υπάρχει ένα άλλο κέντρο επιχειρήσεων σε απόσταση ενός μιλίου που ασχολείται μονάχα με ανθρωπιστικά θέματα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες για την ανάπτυξη δυνάμεων εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών είναι ουσιαστικά αυτό η υποχρέωση και αρμοδιότητα μάλλον της USAID τα κράτη-μέλη τώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτά που είναι οργανωμένα, πιο, σε πιο προχωρημένο τρόπο, έχουν ένα, μια αίθουσα κρίσης για τα θέματα πολιτικής προστασίας και φυσικών καταστροφών και άλλο για τα πολιτικά και στρατιωτικά θέματα και αυτά τα οποία γίνονται στο ένα επίπεδο έχουν επιρροή σε αυτά που γίνονται στα άλλα. Μπορεί, επάνω χάρη, επί τη βάση της φύσης μιας κρίσης, η πολιτική η ομάδα κρίση για την πολιτική προστασία θα ακούσει και την άποψη των εξωτερικών υποθέσεων. Λοιπόν, συμφωνώ ότι χρειαζόμαστε περισσότερη εκπαίδευση, ιδίω για αυτού που είναι πολύ σημαντικοί για μα, του στρατιωτικού, του εργαζόμενου στην ανάπτυξη. Αλλά τόσο μας έχουν ξεπεράσει οι κρίσεις που τα έχει στο προσωπικό μου και εγώ η ίδια. Υπάρχουν κάποιες στιγμές τη μέρα, η οποία έχει όπως ξέρετε μόνο 24 ώρες και στη βδομάδα που έχει μόνο 7 εβδομάδες, που δεν τα βγάζουμε πέρα. Και γι' αυτό θέτω το θέμα των πόρων. Έχει αλλάξει η εργασία μας, έχει αυξηθεί η συχνότητα των κρίσεων, έχει αυξηθεί η πολυπλοκότητα των κρίσεων. Αν θέλουμε να κάνουμε σωστά τη δουλειά μας πρέπει να το αναγνωρίσουμε. Πρέπει να ξέρουμε ότι είναι πολύ σημαντικό να είμαστε σωστά προετοιμασμένοι. Κάποια πράγματα τα καταφέρνουμε, μπορούμε να κάνουμε περισσότερα. Έχουμε κάνει ήδη για την ευελιξία αρκετά πράγματα, αλλά βέβαια πρέπει να κάνουμε ακόμη περισσότερο. Γιατί αν χάσουμε την ευελιξία μας, άνθρωποι χάνουν τη ζωή τους, γιατί κάθε κρίση είναι και διαφορετική. Όσον αφορά τώρα το εθελοντικό σώμα, Είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί στο πώς προχωρούμε. Θέλουμε να εξασφαλίσουμε ότι ό,τι προτείνουμε πραγματικά καλύπτει ένα κενό και κάνει και καλή δουλειά. Συμφωνώ με την μείωση του κινδύνου των καταστροφών. Είναι μία από τις προτεραιότητές μας, μία από τις νομοθετικές μας προτεραιότητες και ούτως ή άλλως θα υποβάλουμε και σχετική ανακοίνωση για την ετοιμότητα αντιμετώπισης των καταστροφών αυτών. Και πραγματικά με πολύ ενδιαφέρον άκουσα τη σύστασή σας για το τι πρέπει να κάνουμε. Ειδικότερα ε, από τη στιγμή που και ο Επίτροπος Ανάπτυξης και της Ανθρωπιστικής Βοήθησης είναι από καινούργιες χώρες. Από νέες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και πραγματικά ε, έχουμε κάνει πολύ σημαντική προσπάθεια στους τομείς της ανάπτυξης και της ανθρωπιστικής βοήθειας. Τώρα, όσον αφορά την έκφραση των συζητήσεων, και μιλάω για το ερώτημα της κυρίας Κέλλερ για την ε, περίοδο μετά την καταστροφή. Μετά από κάθε μεγάλη καταστροφή προσπαθούμε να κάνουμε έναν απολογισμό και να δούμε τι ακριβώς σημαίνει για μας, τι πρέπει να κάνουμε διαφορετικά. Προσπαθούμε να το συμπεριλάβουμε αυτό στις νομοθετικές μας προτάσεις και την οργάνωση των εργασιών μας. Πολλά από τα μαθήματα που έχουμε μάθει αντικατοπτρίζονται ε, στις ε, ανακοινώσει μας ή στις νομοθετικές μας πρωτοβουλίες. Αν θέλετε τη δική μου προσωπική άποψη τι εγώ θεώρησα ότι ήταν το πιο σημαντικό μάθημα που μάθαμε, είναι ότι όταν έχουμε να αντιμετωπίσουμε μία περίπλοκη κρίση και οι συνθήκες είναι δύσκολες, πρέπει να υπάρχει συντονισμός με τα κράτη-μέλη. Η Ευρώπη πρέπει να ε, αναλαμβάνει δράση με ενιαίο τρόπο δεν υπάρχει λόγος ούτε να επικρίνουμε τα ε, Ηνωμένα Έθνη, ούτε άλλες χώρες, αν δεν μπορούμε εμείς μεταξύ μας να συντονιστούμε. Είναι απολύτως απαραίτητος ο συντονισμός. Δεύτερον, πρέπει πάντοτε να προσπαθούμε να βλέπουμε ποιοι είναι οι Ποιε είναι οι πιο ευαίσθητε ομάδε, οι πιο ευάλωτε ομάδε, γιατί ενδεχομένω να μην είναι ε, ισχυρότερη φωνή, να μην ισχυρή η φωνή του. Είναι λοιπόν πάρα πολύ δύσκολο να αντιμετωπίσουμε, να εντοπίσουμε για παράδειγμα, στη Δυτική Όχη, όχι 62% της περιοχής ε, δεν έχει λάβει ιδιαίτερη προσοχή και εκεί είναι οι περισσότερο ευάλωτοι άνθρωποι, η κοινότητα των Βεδουίνων. Ε, είναι λοιπόν, πρέπει λοιπόν να εξασφαλίσουμε εμείς ως Ευρωπαίοι ότι ανταποκρινόμαστε σε, αυτή, σε αυτό το στόχο ε, Τη ανακούφιση των πιο ευάλωτων πληθυσμών και δεν έχουν και κανέναν άλλον άνθρωπο να μιλήσει εκ μέρου τους ε, στο υψηλότερο πολιτικό επίπεδο και πρέπει να το κάνουμε εμείς αυτό. Και κάτι ακόμη το οποίο έμαθα ε, από το περασμένο έτος, ε, όσο περίεργο, όσο κοινότοπο και αν ακούγεται, είναι ότι πρέπει να περιμένει κανείς κάτι που είναι εντελώς απίθανο, γιατί μπορεί πράγματι να συμβεί. Δηλαδή, όταν ε, μιλούσα στη Ουάσιγκτον ε, για μια καταστροφή και είπα ας πούμε ότι 14 ε, μήνες στη δουλειά αυτή έχω δει οποιαδήποτε κρίση μπορεί να φανταστεί κανείς με, με, την εξαίρεση ενός κομίτη που, που έπεσε στη γη ας πούμε. Μόνο αυτό δεν έχω δει και μέσα σε 14 μήνες έχω δει τα πάντα, έχουν δει τα μάτια μου τα πάντα. Αυτό έλεγα νομίζεις ότι έχεις δει πάντα τα χειρότερα και μετά εμφανίζεται κάτι ακόμη χειρότερο στην Ιαπωνία για παράδειγμα. Οπότε, συγγνώμη κιόλα, γιατί έχω μακρηγορήσει πάρα πολύ και το καταλαβαίνω και ε, δεν θα πρέπει να είχατε κάνει αυτή την ερώτηση γιατί τελικά ε, είδατε το αποτέλεσμα είναι ότι μιλάω το σύνορα. Το σημαντικό λοιπόν είναι να αναγνωρίσουμε ότι η συνεργασία δεν είναι μονόδρομος οι αναπτυγμένες χώρες ε, δεν είναι οι αναπτυγμένες χώρες που βοηθούν τις αναπτυσσόμενες. Είμαστε σε έναν κόσμο όλοι, πρέπει να υπάρχει συνεργασία αμφίδρομη, δηλαδή πρέπει να συνεργαζόμαστε, τελεία. Έχουν, γίνει, έχουν υπάρξει ε, τεράστιες κρίσεις, Αυστραλία, Νέα Ζηλανδία, Ιαπωνία, ε, Ηνωμένε Πολιτείε και την καλύτερα, την πιο έτοιμη χώρα, την Ιαπωνία, τη γονάτισε αυτή η θεομηνία η Ιαπωνία χρειάστηκε βοήθεια εξωτερική. Δηλαδή αυτό φαινόταν κάτι το εντελώς απίθανο να συμβεί. Όσον αφορά τώρα τη Λιβύη και, τη, τη Λιβύη και την ε, ε, ανάπτυξη στρατιωτικών δυνάμεων, η θέση μας είναι πάρα πολύ σαφής. Ε, η ανθρωπιστική βοήθεια θα εξαρτηθεί από στρατιωτικές δυνάμεις ως ε, τελευταία δυνατή λύση. Αν δηλαδή δεν υπάρχει καμία άλλη λύση στη Λιβύη, εξακολουθούμε να έχουμε κάποια πρόσβαση, αλλά είναι δύσκολα τα πράγματα. Ε, αν χάσουμε την ε, πρόσβασή μας, τότε θα ζητήσουμε από την EU4 να εμπλακεί. Υπάρχουν ε, πολλοί τρόποι να ε, υπάρξει στρατιωτική παρέμβαση, για παράδειγμα στρατιωτικά σκάφη για την εκένωση ε, υπηκών τρίτων χωρών ή τραυματιών, στρατιωτικά αεροσκάφη για ανθρωπιστική βοήθεια στη Λιβύη ή στο Πακιστάν, η μεταφορά ανθρώπων για που ασχολούνται με την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας. Πρέπει λοιπόν να εξασφαλίσουμε και να αναγνωρίσουμε ότι υπάρχει εντολή της EU4 ε, και λέει όχι στρατιωτική μπότα επιτόπου, ε, κάτι το οποίο είναι ένας περιορισμός και σημαίνει ότι πρέπει να αποφύγουμε ε, οποιαδήποτε στρατιωτική ανάπτυξη γιατί ό,τι και να, κάνουν, ε, να κάνει ένα στρατιωτικό σώμα τι θα κάνει ας πούμε στη Μισράτα αν δεν, υπάρχουν, ε, αν δεν υπάρχει επαρκής ασφάλεια πώς, πώς μπορούμε δηλαδή να ασφαλίσουμε μια πόλη σαν τη Μισράτα Γι' αυτό ακριβώς ε, είμαστε πάρα πολύ ευγνώμονες ότι τα Ηνωμένα Έθνη ομοφόνως ενέκριναν το ψήφισμα που λέει, που, που λέει ότι πρέπει να ε, σώσουμε τους ανθρώπους στη Βεγγάζη. Είμαστε ευγνώμονες γι' αυτό. Αλλά πρέπει να κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για να βοηθήσουμε χωρίς να καταφύγουμε στην ε, στρατιωτική βία. Και για την τελευταία ερώτηση μάλλον δεν την κατάλαβα καλά. Ίσως μετά τη συνεδρίαση αν θέλετε διμερώς να σας την απαντήσω ή δεν ξέρω θέλετε να την ξαναθέσετε τώρα ή να μου την εξηγήσετε. Για την συνάντηση στο Βουσάν και την αποτελεσματικότητα της βοήθειας. Τι πιστεύετε πρέπει να γίνει από την άποψη της ανθρωπιστικής βοήθειας. Εδώ Υπάρχουν δύο σκοπιέ από τι οποίε πρέπει να δούμε την αποτελεσματικότητα. Πρώτα απ' όλα το κατά πόσον θα έχουμε πολλαπλά όργανα, γιατί εδώ έχουμε και με κυβερνητικέ οργανώσει και ε, φορεί του ΟΗΕ και πώ μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα καλύτερο περιβάλλον για την καλή συνεργασία όλων αυτών και την αποφυγή των επικαλύψεων, των επαναλήψεων. Να μην κάνουν πολλοί φορεί τα ίδια Κάτι άλλο που είναι πολύ σημαντικό για μας είναι το πώς θα αυξήσουμε τα αποτελέσματά μας έχοντας και περισσότερο εύστοχα αποτελέσματα. Και όλα αυτά πάντοτε με τη λογοδοσία. Χρειάζεται πάντοτε περισσότερο και περισσότεροι και περισσότεροι. Και όπως είπα, ξοδέψαμε 1,1 δις ευρώ πέρσι δώσαμε σε 140 εκατομμύρια ανθρώπους ε, τρόφιμα, στέγη, ε, ανθρωπιστική βοήθεια, φάρμακα, ό,τι χρειαζόταν. Όσο περισσότερο καλύψουμε, τόσο περισσότερα αποτελεσματικοί θα είμαστε. Το θέμα του συντονισμού λοιπόν θα μας απασχολήσει και από την πλευρά της ανθρωπιστικής βοήθειας. Ευχαριστούμε, ο κύριος Γκέρενς. Ευχαριστώ. Καταρχάς, θα έπρεπε να πω ότι είναι πολύ αποτελεσματική υπηρεσία της κυρίας Γεώργιεβα. Είστε πολύ παρούσα, ε, ιδιαίτερα ενεργή στο ρόλο σας. Αλλά το ερώτημα μου πάει λίγο παραπέρα. Έτσι όπως έχουν τα πράγματα, πρέπει να δείξετε ότι μπορείτε να αντιδράσετε άμεσα στις προκλήσεις. Διότι οι καταστροφές προφανώς δεν είναι προβλέψιμες. Όμως, εγώ θέλω να μιλήσουμε για καταστροφές που μπορούν να προβλεφθούν. ίσως και μακροπρόθεσμα. Μιλώ για τον προβληματισμό που υπάρχει σχετικά με, την, ε, με το λοιμό. Ποια θα ήταν η προστεθέμενη αξία της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε αυτό το σημείο. Ας δούμε τη Δυτική Αφρική ως παράδειγμα. Νομίζω ότι το θέμα της επισητιστικής ασφάλειας εδώ είναι κάτι που δεν μπορεί να καλυφθεί σε περιφερειακό επίπεδο. Στην, στον είναι υπάρχει σοδιά που να φτάνει για να καλυφθούν οι τροφικές ανάγκες του πληθυσμού με την Ιγυρία που έχει μεγάλη αγοραστική δύναμη μπορεί χάρη στις συμφωνίες ελεύθερων συναλλαγών μεταξύ των δύο χωρών αυτών να εξαχθούν προϊόντα ενώ δεν θα καλύπτει τις δικές του τοπικές ανάγκες. Εδώ λοιπόν θεωρητικά υπάρχει κάλυψη των επιστημιστικών αναγκών, όμως τα αποθέματα μακροπρόθεσμα δεν καλύπτουν αυτές τις ανάγκες τις τοπικές, αλλά τις εμπορικές. πριν οι πρώτοι επικαιοκράτες φτάσουν σε αυτήν την ε, Ήπειρο, οι κάτοικοι της περιοχής Νοτιού της Σαχάρας είχαν πολιτική αποθήκευση των τροφίμων, στρατηγική αποθήκευση των τροφίμων. Και προέβλεπαν ότι μπορεί να υπάρξει τριετία ξηρασίας μετά την αποθήκευση. Αυτό είναι ένας τρόπος να αντιμετωπιστεί οποιασδήποτε μορφής ε, επισητιστική καταστροφή. Εδώ λοιπόν αυτό σε εθνικό επίπεδο δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί. Θα πρέπει να γίνει αυτό σε περιφερειακό επίπεδο τουλάχιστον. Και επειδή η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ο μόνο παραγόν, ίσω η Γαλλία, η Γερμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο να μπορούσαν να καλύψουν κι άλλε περιοχέ. Όμω η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πραγματικά ο μόνο διεθνή φορέα που θα μπορούσε να παρέμβει σε, σε περιφερειακό επίπεδο. Τι θα κάνετε εσείς για αυτό το σκοπό. Δεν χρειάζεται εδώ μια στρατηγική εταιρική σχέση. Δεν πρέπει να υπάρξει επισητιστική συμφωνία στο επίπεδο αυτή τη γεωγραφική ζώνη που να γίνει αποδεκτή από τι 15, 16, 17 χώρε αυτή τη περιοχή. Γιατί αλλιώ η αντίδραση μπορεί να είναι αρκετά απότομη. Εάν δεν γίνουν αποδεκτές ε, αυτές οι προϋποθέσεις, ε, για την πρόληψη των επικείμενων ε, καταστροφών θα πρέπει όσοι αρνηθούν τη συμφωνία να αναλάβουν και τις ευθύνε του. Σήμερα εγώ δεν έχω απάντηση. Ξέρω ότι είναι ιδιαίτερα ευαίσθητο το θέμα. Όμως η πρότασή μου είναι η εξής. Δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε μια προσωμείωση και μεταξύ της δικής σας υπηρεσίας και της υπηρεσίας του κυρίου Πίμπαλξ και του κυρίου Ντεχούχτ να δούμε τι μπορεί να γίνει επιπλέον σε αυτό το τομέα. Δεν λέμε ότι θα προβλέψουμε όλες τις καταστροφές, αλλά ίσως να είμαστε προετοιμασμένοι για κάποιες από αυτές. Καμία προβολή δεν... Μάλλον καμία προβολή δεν θα υπάρξει για όλα αυτά, γιατί τέτοιες καταστροφές δεν πρόκειται να μπουν στις ειδήσει των 8. Όμως, δεν μπορούμε να δούμε το θέμα και από αυτή την σκοπιά. Να σκεφτούμε στρατηγικές εταιρικέ σχέσεις και στην επόμενη συνάντησή μας να έχουμε ετοιμάσει και ένα σχετικό έγγραφο ώστε να συνδυαστούν οι ερμηνείε τη δική σα υπηρεσία, τη υπηρεσία του κ. Πίμπαλξ και των ε, κρατών εταίρων μα. Πρόταση ή σχόλιο ήταν αυτό, αν θέλετε, μεθοδολογικού χαρακτήρα, περισσότερο από ό,τι ερώτημα. Πολύ καλή ιδέα σα, αν μου επιτρέπετε, λέει η κυρία Στίφλερ. Θα δώσω το λόγο και στην κυρία Θεοχάρου τώρα. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Κυρία Επίτροπε, εκτιμώ πάρα πολύ την δουλειά που κάνετε και την πολιτική, φιλοσοφική προσέγγιση που έχετε για αυτά τα ζητήματα. Συμφωνούμε σε πολλά ζητήματα. Συμφωνώ και στο γεγονός ότι η πολιτικοποίηση είναι ο μεγαλύτερος κίνδυνος στην παροχή της ανθρωπιστικής βοήθειας. Βεβαίως θα διαφωνήσω μαζί σας για το παράδειγμα που δώσατε όσον αφορά τον κύριο Σάμα, τον Μπαρακ που παρακολουθούσε την εκτέλεση του Οσάμα Μπιλάτεν Εκείνο το άλλο γραφείο που είπατε που ήταν πάρα πέρα και έβλεπε την ανθρωπιστική σκοπιά, το μόνο που με έκανε να σκεφτώ ήταν πώς να το πλύνουν το πτώμα, να το δηλήξουν στη σενδόνη, την καθαρά και να το ρίξουν στη θάλασσα. Καταλαβαίνετε ότι ήταν λίγο, λίγο σκληρό. Βεβαίως παράλληλα θυμήθηκα κυρία Επίτροπε και τον προσιλητισμό, δηλαδή όλο αυτό το θέμα που γινόταν τόσα χρόνια, να δίνουμε την βίβλο στους Αφρικανούς και στη συνέχεια να τους παίρνω με τη γη. Θυμήθηκα, μου φαίνεται ότι το είπε ένας Αφρικανός ηγέτης, νομίζω ότι ήταν ο γιο μου Κενιάτα, είπε όταν ήρθατε εδώ, κρατούσατε τη βίβλο και εμείς είχαμε τη γη μας, όταν πέρασαν τα χρόνια εσείς είχατε τη γη και εμείς είχαμε την βίβλο. Δεν πρέπει σε καμιά περίπτωση η ανθρωπιστική βοήθεια να χρησιμοποιηθεί και δυστυχώ χρησιμοποιείται σε πολλούς τομείς. Γι' αυτό απαιτείται ένας ανεξάρτητος μηχανισμός όπως έχει εισηγηθεί και η κυρία Στρίφλερ, που να παρέχει την ανθρωπιστική βοήθεια σε περιόδους κρίσεως τουλάχιστον, όχι στις χρόνιες καταστάσεις του λοιμού και προβλέψιμες κατά κάποιον τρόπο ε, περιπτώσεις. Άρα είναι, είναι πολύ επικίνδυνο η πολιτικοποίηση της ανθρωπιστικής βοήθειας. Απ' την άλλη όμως και το να ακυρώνεται η ανθρωπιστική παρέμβαση ενός κράτους όπως είναι η Κύπρος ή να προσπαθεί κάποιος να τη μειώσει ή να αφισβητεί την συνέπεια ενός κράτους είναι εξίσου επικίνδυνο. Και αυτό γίνεται πάλι για πολιτικούς λόγους. Έχει γίνει σε αυτή την αίθουσα νομίζω από την α, φίλη την Φρανσέσκα. Ε, δεν μπορεί να αφισβητείτε γιατί δεν μας αρέσει ένα, ένα κράτος ή γιατί δεν μας αρέσει η κατάσταση. Η Κύπρος είναι ένα κράτος κατεχόμενο και αυτό που κάνει είναι από το ιστέρημα της. Και το κάνει γιατί έτσι αισθάνεται ότι πρέπει να κάνει. Ευχαριστώ. Merci Σας ευχαριστώ. Και πάλι ο λόγος στην κυρία Τζόρτζεβα. Να απαντήσετε δύο ερωτήματα, γιατί δεν νομίζω ότι υπάρχουν άλλα ερωτήματα. δέχομαι την ε, πρόσκληση του κύριου Γιώργης να επανέλθουμε για το θέμα αυτό. Κάνουμε κάποια πράγματα, δεν είναι αρκετά. Εργαζόμαστε μαζί με το Παγκόσμιο Πρόγραμμα Διατροφής για να βρούμε τους τρόπους με τους οποίους μπορούμε να βοηθήσουμε τις φτωχότερες χώρες να συνδυάσουν την αγοραστική τους δύναμη και να έχουν μεγαλύτερη επιρροή στις αγορές. <clears throat> Θεωρούμε δεν πρέπει να υπάρχουν καθόλου περιορισμοί για τις ανθρωπιστικές εξαγωγές. Δεν συμφωνούμε για τη Ρωσία που θέλει να θέσει φρένα στις εξαγωγές της. Να το κάνει αλλά όχι για ανθρωπιστικά προϊόντα. Κάναμε λοιπόν κάποια πρώτα βήματα πέρσι που υπήρχε κίνδυνος πραγματικού λοιμού στη Λιποσαχάρια Αφρική, <clears throat> Νίγηρα, Μαλή και Βόρεια Νιγηρία. Είναι μια καταστροφή που δεν έγινε ορατή γιατί ήταν ο σκύλος που όπως την ιστορία του Sherlock δεν γάβησε. Ήμασταν έτοιμοι για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε αυτήν την επερχόμενη καταστροφή. Έχετε δίκιο όμως να το βλέπετε από πολλαπλές οπτικές γωνίες. Έχουμε ξεκινήσει κάποια προσπάθεια για το πώς μπορούμε να εξασφαλίσουμε την ε, επισητιστική ασφάλεια μαζί με τον κύριο Πίμπαλξ και τον Επίτροπο Γεωργίας. Και έχετε απόλυτο δίκαιο ότι Πρέπει και ο κύριος Ντεχούχτ να εμπλακεί σε αυτό το εγχείρημα. Θα ξανασκεφτούμε λοιπόν όλα αυτά τα θέματα και θα επανέλθουμε. Το παράδειγμα με τον κύριο Ομπάμα, ο οποίος παρακολουθούσε από την τηλεόραση ίσως, έρχεται σε επίρρωση όλων αυτών τα οποία λέμε. Είναι γεγονός ότι υπάρχουν και στρατιωτικές και πολιτικές δράσεις <clears throat> και υπάρχουν και ανθρωπιστικές δράσεις, αλλά δεν πρέπει να συγχέονται, δεν πρέπει να ταυτίζονται απόλυτα. Είμαι υπερήφανη γιατί η Κομισιόν πήρε την απόφαση να θέσει τον κύριο Πίμπαλξ και εμένα σε, αυτό το, σε αυτές τις αρμοδιότητες. Εμείς έχουμε μια απουσία απικιακού παρελθόντος και γι' αυτό μπορούμε να είμαστε πιο αντικειμενικοί ίσως. Και αυτό μας δίνει και μια διαφορετική εικόνα όταν εργαζόμαστε σε μέρη όπου το παρελθόν το απικιακό δεν είναι και τόσο φωτεινό. <clears throat> Καταλαβαίνω λοιπόν ότι αυτό το οποίο θέλετε να πείτε είναι ότι αν θέλουμε να μας πάρουν σοβαρά δεν αρκεί το να κινητοποιούμε χρήματα, να έχουμε το σωστό κόσμο, θα πρέπει να υπάρχει και μια θέση επί των αρχών και θα πρέπει να είμαστε ε, να έχουμε σεβασμό για τις αρχές μας και αυτό ακριβώς είναι αυτό που θέλουμε να κάνουμε εμείς. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Στίφλερ. Η επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής μας θα λάβει χώρα στις Βρυξέλλες στις 14 Ιουνίου από τις 3 έως τις 5.30 και την Τετάρτη 15 Ιουνίου από τις 9 στο 10.30 και από τις 3 ως τις 6.30. Μερσή κυρία Επίτροπε που ήρθατε για τη συνεδρίασή μας. Πάντα ερχόσαστε με μεγάλη ορμητικότητα και ενθουσιασμό. Ευχαριστούμε κυρία Γεώργιεβα για την επικοδομητικότητά σας και θα τα ξαναπούμε. Alors, euh, cette se termine. Τελείωσε λοιπόν η συνεδρίασή μας, αλλά θα συνεχίσουμε στο Wicklow στην αίθουσά μας για μια ανταλλαγή απόψεων με την κυρία Μαλόουν της Γενικής Διεύθυνσης ΕΚΟ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την επαναδιαπραγμάτευση της Σύμβασης του 1999 για την επιστηστική βοήθεια και ακολουθούν οι συντονιστές. Σας ευχαριστώ που θα αποχωρήσετε ηρέμος και ησύχως. Για αυτό το σημείο οι μόνοι οποίοι μπορεί να είναι παρόντες είναι οι βουλευτές, οι συνεργάτες τους, το προσωπικό των πολιτικών ομάδων και η Γενική Γραμματεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου εξάλλου, ακόμα και της Κομισιόν. Παρακαλώ τα άτομα τα οποία είναι ξένα προς το λειτουργήμα αυτό να αποχωρήσουν εν σιωπή και ησυχία για να συνεχίσουμε τις εργασίες μας. Ευχαριστώ